για την ε, διορισμό στις ε, αντιπροσωπείες, στις δικνευριστικές αντιπροσωπείες. Αυτά ε, θα αναφέρουμε στα πρακτικά. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι ο συνάδελφος Αντέου Σιμάνσκι, Γιάτσεκ Όλγκερ Γιάτσεκ Γλωτζόβιτς, Σβίλνιεφ από την EFD ε από τις 29 ε, Δεκεμβρίου έχουν προσχωρήσει στο Κοινοβούλιο. Να σας ανακοινώσω επίσης ότι βάσει του άρθρου